<laughs> Καλημέρα σας κυρία Επίτροπε, καλημέρα σε όλους. Άρχεται η συνεδρίαση. Θέμα πρώτον, δήλωση της Επιτροπής με ένα έτος πρακτικής εφαρμογής πρωτοβουλίας των Ευρωπαίων πολιτών. Αξιολόγηση